Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη ψηφοφορία της έκθεσης Λάσλο Σουριάν σε ό,τι αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2010. Άρχεται η ψηφοφορία για την έκθεση Σουριάν. Η ψηφοφορία θα γίνει με ονομαστική κλίση. Παρακαλώ τοποθετήστε τις ε, ηλεκτρονικές κάρτες. Otwieram głosowanie. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Δεκτή έκθεση. Συγχαρητήρια κύριε Σουριάν. Έκθεση Αρία Ετσεβερία. με θέμα την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου. Ψηφίζουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παρακαλώ, κύριος Πόσελτ. Διαδικαστικό. Κοίταξε την κάρτα μου, την ξέχασα στην Επιτροπή Εξωτερικών Πολιτικών Υποθέσεων. Μου τη φέρνουν. Ε, και εγώ ήμουν εδώ από την πρώτη ψηφορία. Ε, δεν μπόρεσα μόνο να ψηφίσω. Απλά ήθελα να το πω. Okay. Okay. You must help it in any way. Ε, Βοηθήστε το παρακαλώ θα ψηφίσουμε την έκθεση Αρία Ετσεβερία για την ολοκλήρωση τη εσωτερική αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου. Ζα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Ε, Συγχαρητήρια κύριε Ετσεβερία. Ψηφίσουμε τώρα την έκθεση Κριστίν Τεβεϊράκ με θέμα την διερεύνηση και πρόληψη αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων. Ψηφίζουμε τις συμβεστικές λύσεις. Συμβαστική λύση πρώτη. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτό. Ψηφίζουμε τώρα την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Με ονομαστική ψηφοφορία Άρχιτε ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Συγχαρητήρια, κυρία Ντεβεϊράκ. Ο κύριος Τσουκάλας ζήτησε το λόγο. My, my, my card is not... Δεν δούλεψε η κάρτα μου κύριε. Για τις προηγούμενες δύο ψηφοφορίες έγινε αυτό. Δεν δουλεύει. Ούτε λειτουργεί. Παρακαλώ να στείλουμε τεχνικό στην έδρα 831. Σας ευχαριστώ για την ε, πληροφορία κύριε Τσουκαλά. Περνούμε στην έκθεση του κυρίου Βιντάλ Κουάδρας για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο. Πρώτο μπλοκ, συμβαστική λύση. Ποιος είναι υπέρ της πρώτης συμβαστικής πρότασης. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροποποιημένη πρόταση επιτροπής. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Θερμά συγχαρητήρια κύριε Βιντάλ Κουάδρας. Ο κύριος Σόγκορ ζήτησε το λόγο, που είναι άλλωστε και ο εισηγητής της επόμενης σύστασης. Παρακαλώ, είμαι υπέρ. Ο κύριος Λαντσμπέργης μιλάει, όχι ο κύριος Σόγκορ. Είμαι υπέρ. Καλώ θα το δούμε αργότερα, κύριε Ευρωβουλευτά. Ο κύριος Σόγκορ ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δήλωση που έκανε. Εδώ πρόκειται για την επανεισδοχή, για την Συμφωνία Επανεισδοχής με το Πακιστάν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε τη σύσταση για τη Συμφωνία Επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακιστάν. Δεν κατατέθηκαν τροπολογίε. Θα ψηφίσουμε ε, το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. Καλώ. Θα γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση της προηγούμενης ψηφοφορίας. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Συγχαρητήρια κύριε Σόγκορ. Επόμενο θέμα, η έκθεση με την Καζάκ για τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία. Σχέδιο ψηφίσματος. Διαδικαστικό. Ο κύριος Στογιάνοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το άρθρο 175 θα ήθελα να επικαλεστώ και να ζητήσω αναπομπή της έκθεσης αυτής στην αρμόδια επιτροπή. Ο κύριος Καζάκ αντιμετωπίζει σύγκρουση αρμοδιοτήτων, ε, ασυμβίβαστο μάλλον, γιατί ε, χρηματοδοτήθηκε από την ε, τουρκική κυβέρνηση για να ε, κάνει τι ανώτερε σπουδέ στη Σορβόνη. Δεν είναι καθόλου αντικειμενικό και αμερόληπτο λοιπόν σε ό,τι αφορά την έκθεσή του. Επίση, θα ήθελα να προτείνω τον διορισμό νέου εισηγητή που θα είναι πιο αντικειμενικό και αμερόληπτο και ελπίζω ότι θα με υποστηρίξουν οι συνάδελφοι σε αυτό το αίτημα. Τέτοιου είδου αιτήματα μόνο μια πολιτική ομάδα δικαιούται να τα υποβάλει. Ε, είναι μη παραδεκτό το αίτημά σα, δεν μπορούμε καν να το εξετάσουμε θα περάσουμε στην ψηφοφορία της έκθεσης Καζάκ για τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 1. Ονομαστική κλίση. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 2. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το σημείο 2, κύριε Πρόεδρε, προβλέπει ε, είτε μια πολιτική ομάδα, τουλάχιστον 40 ευρωβουλευτές ε, μπορούν να ζητήσουν αναπομπή μιας έκθεσης στην αρμόδια επιτροπή. Παρακαλώ να ρωτήσετε την, ε, την Ομίγυρη, αν υπάρχουν 40 ευρωβουλευτές που είναι υπέρ του αιτήματο του δικού μου. Υπάρχουν, λέει ο πρόεδρος, ψήφοι υπέρ του αιτήματο στο Γιάννοφ. Δεν αρκούν ε, οι βουλευτέ που σηκώθηκαν για να υποστηρίξουν το αίτημά σα, ε, κύριε Στογιάννοφ. Δεν συγκεντρώνεται τον αριθμό των 40 που απαιτείται από το σχετικό εδάφιο. Ανεπαρκής αυτή η πλειοψηφία. Επανερχόμαστε λοιπόν. Σα υπενθυμίζω ότι ψηφίσαμε υπέρ του πρώτου τμήματος της τροπολογία 2. Θα περάσουμε στο δεύτερο τμήμα. Ποιο είναι υπέρ. Δεύτερο τμήμα της τροπολογία 2. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Για το τμήμα 2 της τροπολογίας 2. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του ψηφίσματος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Καζάκ. Επόμενη έκθεση της κυρίας Δελάνκε με θέμα την ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό τη διατήρηση της βιοπικιλότητας. Ψηφίζουμε την παράγραφο 51. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η εισηγήτρια. Έχετε το λόγο κυρία Ντελάγκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλά να σας ζητήσω ε, να ψηφίσουμε ε, για το τελική ψηφορία για το ψήφισμα να είναι ονομαστική. Το έτοιμά σας ε, καλύπτεται από πολιτική ομάδα. Εκ μέρους πολιτικής ομάδας υποβάλλεται αυτό το αίτημα. Προφανώς συζητήθηκε και με τους και ηγητές. Προφανώς. Ευχαριστώ. Um, Κοιτάξτε, λίγο καθυστερημένα ε, θέσατε το αίτημα αυτό, αλλά αν δεν διαφωνεί κανείς, να ψηφίσουμε με ονομαστική ψηφορία. Υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί. Εσείς διαφωνείτε. Μάλιστα, εγώ διαφωνώ, όχι γιατί είμαι κατά της ονομαστικής ψηφοφορίας, αλλά το έχω πει επανειλημμένα εδώ. Ε, θα πρέπει να έχουμε τους ίδιους κανόνες ε, για όλα. Ε, όταν εγώ ζήτησα ονομαστική ψηφοφορία για κάτι άλλο, μου τα απορρίψατε. Αν λοιπόν υπάρχουν κανόνες, να τηρούμε τους κανόνες. Πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, 60 7 ξεχωριστή ψηφοφορία ε, ποιος είναι παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο κομμάτι ποιος είναι υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται το 69 ξεχωριστή ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα ε, υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε για το σύνολο του ψηφίσματος. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Κύριε Πρόεδρε, με κάθε σεβασμό θα ήθελα να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε αυτή τη διαδικασία. Μπορούμε και κατά τη διάρκεια τη ψηφοφορία να ζητήσουμε ονομαστική ψηφοφορία. Και αν 40 βουλευτέ είναι κατά, καταρρύπτεται το, το αίτημα. Αλλά μόνο ένα ευρωβουλευτή δεν είναι κατά το αιτήματο ονομαστική ψηφοφορία. Θα ήθελα, παρακαλώ, ψύχρεμα, να διευκρινίσω το εξή. Η διαδικασία που επικαλεστήκατε αφορά τις προφορικές τροπολογίες. Για τις προφορικές τροπολογίες δεν ισχύει η προθεσμία. Αν προτείνετε ψηφοφορία με ονομαστική κλίση, αν προτείνετε λοιπόν ονομαστική ψηφοφορία, ε, τότε ισχύει άλλο θέμα. Κανένας δεν μπορεί να αντιταχθεί. Αλλά υπήρχε μία προθεσμία και εσείς δεν την υποβάλλατε εμπρόθεσμα αυτή την αίτησή σας. Αυτό προβλέπει ο κανονισμός. Το αίτημά σας είναι εκπρόθεσμο. Γιατί για τέτοιου είδους αιτήματα ισχύει η προθεσμία. Από τη στιγμή που ισχύει η προθεσμία, κανείς δεν μπορεί να αντιταχθεί. Εγκρίθηκε το ψήφισμα. Σε χαρητήρια, κυρία Δελάγκε για την προσπάθειά σας και το έργο σας. Προχωρούμε στην επόμενη ψηφοφορία της έκθεσης Φεραίρα. We were voting, colleagues. Συνάδελφοι, παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πόσες φορές να ψηφίσουμε, δηλαδή. Μία. Ψηφίσαμε και ήταν σαφές το αποτέλεσμα. Σαφέστατο. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με την έκθεση Φερέρα με θέμα την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έχουν καταθέσει τροπολογίες. Ψηφίζουμε το σχέδιο ψηφίσματος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μπράβο σας κύριε Φερέιρα. Παρακαλώ, έκθεση Θεοχάρου τώρα, μείωση τη φτώχεια και δημιουργία απασχόληση σε αναπτυσσόμενε χώρε. Δεν έχουν κατατεθεί τροπολογίε. Σχέδιο ψηφίσματο. Θα ψηφίσουμε χωριστά τι παραγράφου. Δεύτερη παράγραφος, ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 26. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 49. Ποιος είναι υπέρ. Ε, 26. Παράγραφος 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αλλά σωστά ζητήσατε επαλήθευση. Σας ευχαριστώ που το επισημάνατε. Γιατί είχαμε την αίσθηση ότι ήταν μεγαλύτερη διαφορά. Παράγραφο 49. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 54. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 83. Ψηφοφορία κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται. Παράγραφος 84. Η κυρία Θεοχάρου ζήτησε το λόγο. Προφορική τροπολογία για την παράγραφο 84. Έχετε το λόγο κυρία Θεοχάρου. Προφορική τροπολογία η οποία είναι ως ακολούθως I will read the English θα διαβάσω το αγγλικό κείμενο. Καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ομάδα G20 να λάβουν συγκεκριμένες ενέργειες ε, για να καταργήσουν ε, την φοροδιαφυγή, τους φορολογικούς ε, παραδείσους από διάφορες χώρες και να προάγουν το να επενδυθούν οι πόροι αυτοί στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και μετά τις τρεις πρώτες λέξεις έχουμε το G20 και εδώ γίνεται την κατάσταση με το ρήμα προ Υπάρχουν αντιρρήσεις, γιατί θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι θα πρέπει 40 να είναι κατά για να απορριφθεί το αίτημα προφορική τροπολογία. Δεν υπάρχουν αντιρρήσει, οπότε ψηφίζουμε μαζί την προφορική τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ για την παράγραφο 84, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφο 94, Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για την παράγραφο 94. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Για το 21 ε, θεωρώντας ποιος είναι υπέρ. Κατά. Μάλλον απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται το 21. Αιτιολογική σκέψη Β. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. αποχές απορρίπτεται. Το σύνολο του νομοθετικού ψηφίσματος, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Θεοχάρους. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Όταν επιστρέψετε θα βρείτε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο κάποιες πληροφορίες που σας στείλαμε για την Πέμπτη. Το επαναλαμβάνει και αγγλικά ο πρόεδρος. Σας στείλαμε mail με πληροφορίες για την Πέμπτη. Παρακαλώ, ελέγξτε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. Well, I would like to speak to the lady 583.

start the explanation of votes. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Αρίας Εσεβέρια θα πάρει το λόγο ο κύριος Μεσ...